Επανάληψη τη Συνόδου, τα πρακτικά τη χθεσινή της χθεσινής τα έχετε στη διαθεσή σας, δεν ξέρω αν υπάρχουν ενστάσεις, όχι μάλιστα, άρα τα πρακτικά εγκρίνονται. Από το Συμβούλιο σε πρώτη ανάγνωση και την